Εδώ πέρα χρειαζόμαστε ευρεία συνένεση, οπότε θα ήθελα να πω το εξής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις συζητητές στη Γραμματεία για, για το εξαιρετικό τους ε, έργο. Σήμερα δεν έχουμε ακόμα καταλήξει ένα οριστικό αποτέλεσμα. Αποζημίωση των επενδυτών ε, για όλα τα πιθανά ε, αξιόγραφα. Όσο ε, πελάτης, ως πενητής μπορεί κανείς να αποζημιωθεί από το κράτος ε, σε περιπτώσεις απάτης και αμέλειας και κακοδικίας. Όχι δηλαδή εάν η επένδυσή του απλά χάσει την αξία της. Τώρα για τις τροπολογίες κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, μιλήσαμε για 100.000 ευρώ ανά επενδυτή ανεξαρτήτως χώρας. Υπάρχουν χώρες που έχουν 100.000, υπάρχουν ε, άλλες που είναι ε, μόνο στις 5.000, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και τα λοιπά. Δεν θέλουμε να μειώσουμε το ε, ποσό και να επιδεινωθεί η κατάσταση σε κάποιες χώρες πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα επενδύουν στο μέλλον των ε, επιχειρήσεων. Θα πρέπει να καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες έχει αποδειχθεί στο δικαστήριο πως υπήρχαν κακές συμβουλές οι οποίες δόθηκαν από επενδυτικές εταιρείες και άρα οδηγήθηκαν κάποιοι σε κακές επενδυτικές ε, αποφάσεις. Ε, π.χ. Ε, σύμβουλοι οι οποίοι συμβολεύουν ηλικιωμένους να επενδύσουν σε πολύ επικίνδυνα κοινά ταμεία και επενδυτικά προϊόντα. Οπότε δεν θα πρέπει εδώ πέρα να υπομειστεί το βάρο ο φορολογούμενο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ταμείο εξάντε το οποίο θα χρηματοδοτούν οι εταιρείε για την περίπτωση χρεοκοπία και θα πρέπει να είναι από 0,5 έω 0,3% της ε, αξίας ε, των ε, αξιογράφων που διαχειρίζονται και βεβαίως να περάσουμε από την δεκαετία στην πενταετία και βεβαίω θα πρέπει μεγαλύτερε επιχειρήσει να συνεισφέρουν περισσότερο και ειδικά αυτές οι οποίες αναλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους. Τέταρτον, πρέπει και ο δανειοδοτικός μηχανισμός να ε, προσαρμοστεί. Η Κομισιόν θέλει ένα σύστημα υποχρεωτικό που όλοι θα μπορούν να δανείζονται για να μην υπάρχει ηθικός κίνδυνο και να μην υπάρχει υποχρηματοδότηση. Προτείνουμε λοιπόν να μην ε, λειτουργήσει μέχρι να έχουν φτιάξει όλα τα συστήματα, τα ταμεία τους και μετά από μία πενταετία θα πρέπει να είναι δυνατός ο δανεισμός υπό τον όρο τα συστήματα αυτά να έχουν φτάσει τον ε, στόχο, το επίπεδο του στόχου. Πέμπτον, η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει τι γίνεται με τα ΟΣΕΚΑ το εάν θα πρέπει να συμπεριληφθούν ή όχι. Θεωρούν πως πρέπει να το ξαναδούμε αυτό για να δούμε πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει. Μην ε, έχουμε άλλα σκάνδαλα τύπου Μάντοφ. Ε, θεωρούμε πως η Κομισιόν θα πρέπει να το ε, δει αυτό το θέμα και πιθανώς ε, να το επεκτείνει με περαιτέρω ασφάλιση. Και επιπλέον βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, να υπάρχει μια υποχρέωση να ενημερώνονται τα κρατημέλη, η Κομισιόν και η ΕΣΜΑ. Κύριε Πρόεδρε, η προστασία των επενδυτών είναι σημαντική για τους επενδυτές και για τη χρηματοδότηση οικονομική σταθερότητα. Χρειάζομαι αύριο σαφή απόφαση του Κοινοβουλίου και ελπίζω να με στηρίξετε για να μπορέσω να πάω διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον Όλε Σμιτ και όλα τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων Πρόκειται πραγματικά για το φιλόδοξο μήνυμα το οποίο δώσατε κύριε Όλε Σμιτ και που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση του συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών. Αυτό είναι ένα, μια ψηφίδα σε ένα συνολικό πλαίσιο που εξασφαλίζει <clears throat> την ασφάλεια των, ε, συμπληρώνει το νομοθέτημα για την ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων και των ασφαλιστικών συμβολέων. Είναι μια σημαντική λοιπόν πρόταση της Κομισιόν για να αντιμετωπίσουμε την κρίση γιατί οι λιανικοί επενδυτές είναι κατά κάποιο τρόπο οι πιο ευάλωτοι στις κρίσεις και ήταν και τα πρώτα θύματα της κρίσης. Δεν πρόκειται μονάχα λοιπόν για το να τους προστατεύσουμε και εκεί δεν θα καταλαβαίνανε οι συμπολίτε μας ότι θα μπορούσαμε να στοχίσουμε εκεί. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα το οποίο θα εξασφαλίσει σε ακραίε καταστάσει, όπω απάτε ή σοβαρά λειτουργικά ασφάλματα να του αποζημιώσει κανεί όταν χάνουν όλε τι επενδύσει του. Οι αποζημιώσει αυτέ λοιπόν συμβάλλουν στην ανάκτηση τη εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και έτσι ευνοούν και τη δημιουργία μια πραγματική ενιαία αγορά για, για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Αυτή είναι η λογική λοιπόν η οποία θα πρέπει να πριτανεύσει μεταξύ των συνομοθετών ώστε να προχωρήσει το θέμα αυτό. Η Κομισιόν ήδη από το 1987 είχε προτείνει και είχε εγκριθεί μια οδηγία για την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών, αλλά πρέπει να την βελτιώσουμε και να την προσαρμόσουμε στις σημερινές συνθήκες. Εγώ υποστηρίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό μια προληπτική πολιτική κοστίζει πολύ περισσότερο η θεραπεία από την πρόληψη σε πολλούς τομείς όπως και η οικολογία αλλά και στην οικονομία. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί προληπτικού χαρακτήρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δημιουργείται αυτό το Ταμείο Εγγύηση από αυτού οι οποίοι προσφέρουν στην αγορά αξιόρθα. Κύριε Σμιτ, εγώ συμμερίζομαι λοιπόν καταρχήν τη φιλόδοξή σα προσέγγιση. Και η συμφωνία του Κοινοβουλίου για την προχρηματοδότηση σε ένα ειδικό ταμείο, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και για μα είναι απαράγραπτη προπόθεση για να είναι αξιόπιστο το σύστημα αυτό. δεν, υπάρχει, δεν έχει νόημα να προβλέπει κανείς μια κάλυψη αυτών των επενδύσεων αν δεν υπάρχει η απαραίτητη πρόβλεψη σε, για τους φορείς αυτούς οι οποίοι πρέπει να δώσουν αποζημίωση. Το να πρέπει να βρουν αυτά τα χρήματα σημαίνει πρόσθετη πίεση σε αυτούς τους φορείς. Επίσης το επίπεδο ε, εγγύησης όπως προτείνεται είναι 100.000 ευρώ. Εμείς έχουμε προτείνει ως Κομισιόν κάτι λιγότερο 50.000 ευρώ γιατί θεωρούμε ότι ο κίνδυνος ο οποίος προέρχεται σε συστημικό επίπεδο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πολύ μικρότερος. Μας φαίνεται μικρότερος από ότι στο τομέα των τραπεζικών καταθέσεων. Γνωρίζουμε όλοι τον πανικό τον τραπεζικό και τους καταθέτες οι οποίοι τρέχαν να βγάλουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες το 2008. Τέλος, χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να διατηρήσει <clears throat> το μηχανισμό του αμοιβαίου δανεισμού μεταξύ ταμείων, γιατί αυτό είναι σημαντικό σε μια πιο εναρμονισμένη ε, οικονομική λογική και όπου υπάρχει και μια κατά κάποιο τρόπο καλύτερη κατανομή των κινδύνων για να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις. Εκεί που έχετε κάποιες ε, διαφορές κύριε Όλη Σμίτα με την πρόταση της Κομισιόν αναφέρατε παραγματικά ότι είναι φυσικό να υπάρξει μια επέκταση αυτού του συστήματος στους ΟΣΕΚΑ. Εσείς θέλετε λοιπόν να εφαρμοστεί και εκεί αυτό το σύστημα. Κατανοώ το ότι θέλετε να υπάρξει μια επανεξέταση μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ. Κύριε Σμιτ, <clears throat> μπορείτε να βασιστείτε στην Κομισιόν να προχωρήσει την αναθεώρηση αυτού του νομοθετήματος. Επίσης, η μείωση της προχρηματοδότησης κατά, από 0,5 σε 0,3% αυτό πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Αλλά άμα θέλετε μια κάλυψη επίπεδου 100.000 ευρώ, αν εσείς μειώσετε την προχρηματοδότηση, αυτό θα θέσει το σύστημα πολύ πιο εύκολα σε συστήκες στρες ή δυσκολιών. Τέλος, έχω κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την τροπολογία που θα έχει σαν στόχο να καλύψει τις λεγόμενες κακές συμβουλές. Εγώ κατανοώ τον στόχο σας, και συμφωνώ. Είναι πλοκά όμως τα χρηματοπιστωτικά θέματα. Υπάρχουν πολλοί αγύρτες οι οποίοι πολλές φορές κοροϊδεύουν τους πιο αφελείς επενδυτές. Αυτό είναι περισσότερο όμως μέσα στα πλαίσια της οδηγίας MIFID για τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία. Και εξάλλου είναι δύσκολο να υπάρξει εφαρμογή <clears throat> αυτής της ρήτρας. Αυτό θα διεύρυνε πάρα πολύ τον αριθμό των περιπτώσεων όπου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Αποζημίωσης χωρίς να προτείνεται συγχρόνως μια αύξηση της χρηματοδότησης. Λοιπόν, ως έχουν τα πράγματα αυτά, κύριε Σμιτ, η ιδέα των κακών συμβουλών θα οδηγήσει σε διαφορετικές ε, ερμηνείες από τη μία χώρα στην άλλη και θα οδηγήσει και πάλι σε κατακαιρματισμό των αγορών και των ρυθμίσεων. Γι' αυτό δυσκολευόμαστε να δεχτούμε την έννοια αυτή στο κείμενό μας. <clears throat> Συνολικά όμως κύριε Σμιτ, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη θαυμάσια εργασία που έχετε κάνει και εσείς και οι συντονιστές και οι ισχυώδεις της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι συμμεριζόμαστε μια κοινή προσέγγιση στο θέμα αυτό για μια λύση η οποία είναι φιλόδοξη, είναι ευρωπαϊκή και το Συμβούλιο πρέπει να το λάβει υπόψη. Αυτό και το μήνυμα το οποίο στέλνετε κι εσείς στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να συμφωνήσουν το ταχύτερο δυνατό για μια γενική προσέγγιση στα θέματα αυτά και βασίζομαι στην Πολωνική Προεδρία να αναπτύξει όλες τις προσπάθειες και να, κάνει, να καταφέρει να πείσει τις άλλες χώρες που δεν είναι ακόμα πεπισμένες για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τους μικροεπενδυτές. Είναι απαραίτητο να έχουμε λοιπόν και υψηλή κάλυψη, <coughs> μια αξιόπιστη προχρηματοδότηση στο Ταμείο Ασφάλειας και μια εύκολη πρόσβαση στην αποζημίωση των μικροεπενδυτών. Αυτό, αυτή είναι και η κατεύθυνσή μας και σας ευχαριστούμε κύριε Σμίτ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Μπόντου για την νομική επιτροπή και για ένα λεπτό. Η λειτουργία των συστημάτων αποζημίωσης των παιδιτών έχει στόχο να βελτιώσει τη, και να ευθυγραμμιστεί με την αγορά χρηματοπιστικών μέσων. Δεν μπορεί να υπάρχει ισοδυναμία αντιμετώπιση μεταξύ των επενδυτών στην κεφαλαία αγορά και των καταθετών σε εμπορικέ τράπεζε. Παρότι οι δύο κατηγορίε πρέπει να προστατεύονται, η προστατεία του, των επενδυτών πρέπει να είναι κυρίω δική του ευθύνη. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι καλή ιδέα να αυξηθεί το όριο στι 100.000 ευρώ, διότι τούτο θα θέσει υποβολικά μεγάλο βάρος στους τοπικούς ε, ε ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα διατηρήσει την τοπολογία, την προσωπική τοπολογία, για την αναβολή του, της εφαρμογής της οδηγίας στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για να τηρηθούν και οι διατάξεις της συνθήκης ε, προσχώρησης. Ευχαριστώ. Για τις πολιτικές ομάδες τώρα. Πρώτος, ο κύριος Κοζές, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, συνάδελφοι, ο στόχο του κειμένου είναι να προστατεύσει του ε, ιδιωτικού επενδυτέ από παράνομε ή απατηλέ ε, ή προβληματικέ ε, πρακτικέ επενδυτικών εταιριών. Το κείμενο έχει στόχο να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μετά από μια κρίση κατά την οποία οι μικροεπενδυτές, όπω είπατε και εσεί, κύριε Επίτροπε, ήταν οι πλέον τρωτοί και τα πρώτα θύματα της κρίσης. Πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι το κείμενο αυτό οργανώνει μια αποζημίωση σε ίστατη βάση. Δεν είναι πρώτη, αλλά ίστατη μορφή αποζημίωσης και γι' αυτό η Επιτροπή μας ομόφωνα υπερψήφισε την έκθεση ζητώντας μια μέγιστη εναρμόνιση των κανόνων και άνοδο του ανώτατου ρίου στα 100.000 ευρώ. Για την ιδιαίτερη περίπτωση του ΝΟΣΕΚΑ, η Επιτροπή κρίνει ότι όχι ότι δεν πρέπει να προληφθούν μέτρα προστασία των επενδυτών εκεί, αλλά ότι αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα που έχουν ε, καλή ε, φήμη έχουν, πρέπει να έχουν δικούς τους ειδικού κανόνες στα πλαίσια της αναθεώρηση τη οδηγίας ΣΟΣΕΚΑ. Γι' αυτό η Επιτροπή ζήτησε από την Επιτροπή της Ένωσης να κάνει μια μελέτη για να εξετάσει τα υπέρ και τα κατά της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της παρούσης οδηγίας και στις ΟΣΕΚΑ. Τώρα, το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει ούτω ώστε αυτό που θα ψηφίσουμε σε πρώτη ανάγνωση, θα ψηφίσουμε και το νομοθετικό ψηφίσμα, να γίνει γρήγορα ένα πραγματικό νομικό κείμενο που θα εφαρμόζεται. Και επαναλαμβάνω, για τους ιδιωτικούς επενδυτές της Ευρώπης δείχνουμε τη σημασία της Ευρώπης που υλοποιείται με μια ισοδύναμη προστασία για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από τη Σοσιαλιστική Ομάδα η κυρία Μπερές για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η αναθεώρηση αυτή της οδηγίας για τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών ακολουθεί δυστυχώς την κρίση και το σκάνδαλο Μάντοφ στις Ηνωμένες Πολιτείες το οποίο κτύπησε κατάμουτρα πάρα πολλούς μικροεπενδυτές στην Ευρώπη. Όπως υπενθυμίσατε επίσης, αυτό γίνεται εν με την μεταρρύθμιση της οδηγίας για τις τραπεζικές, τραπεζικές καταθέσεις και για τις ασφαλιστικές και τα, για τις ασφάλειες. Εμείς έχουμε ζητήσει το, η οροφή να είναι 100.000. Αλλά εφόσον το κάνετε αυτό από 25.000 σε 100.000 για τις τράπεζες, γιατί δεν το κάνετε και για τις επενδύσεις. Θέλουμε οι, ευρωπαϊκοί, οι ευρωπαίοι επενδυτές να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους και να δώσουν και επενδύσεις που είναι χρήσιμες για μακροχρόνιες επενδύσεις. Είπατε ότι οι κακές συμβουλές μας παραπέμπουν στην ε, συμφωνία, στην ε, οδηγία για τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία. Αυτές τις ιδέες θέλουμε εμείς να αναφέρουμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πολύ θετική ιδέα που περιείχε αυτή η οδηγία. Εμείς θέλουμε να αντλήσουμε τις, ε, τις απόρριες αυτής της οδηγίας για τα αναλλακτικά ταμεία και σε αυτήν την περίπτωση. Για τα ΟΣΕΚΑ. Έχουμε πει ότι αυτοί οι οποίοι σήμερα έχουν ΟΣΕΚΑ στη διάθεσή τους βρίσκονται σε πολύ πιο δύσκολη θέση με τους επενδυτές που έχουν επενδύσει σε άλλα συστήματα, ενώ παρόλα αυτά αποτελούν μια προσθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά. Τέλος, θέλω να σας αναφερθώ, να αναφερθώ και στο πώς θα αντιμετωπίσει η οδηγία αυτή και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Το ζητούμε όπως θα πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο θα είναι ένα σύστημα ασφαλιστικού χαρακτήρα και να είναι αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσει το <clears throat> ταμείο το εξάντε. Αυτό θέλετε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες μας δεν θα καταλάβουν να μην πραγματοποιηθεί. Βασιζόμαστε λοιπόν στην πίεση που μπορέσει να ασκήσει η Κομισιόν για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα όπου ορισμένε χώρες στο Συμβούλιο δεν θέλουν να προχωρήσουν αρκετά γρήγορα. Φοβάμαι πως ε, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, οπότε θα ήθελα να τηρείτε το χρόνο ε, αγόρευση. Ο κύριος Γκίκολτ για 1,5 λεπτό από τους ε, πράσινους. Ναι, κύριε Σμιτ, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή συνεργασία και για τη θέση την οποία λάβατε εδώ πέρα. Η μεταρρύθμιση αυτή της προστασίας ε, των επενδυτών είναι αναγκαία για βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών των χρηματαγορών. Είδαμε πάρα πολλά μεγάλα σκάνδαλα το ε, αποτέλεσμα είναι αυτή εδώ πέρα η μεταρρύθμιση. Ευχαριστούμε και την Κομισιόν για την ε, απαιτητική πρόταση την οποία υπέβαλε. Σύντομα τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία τα οποία δεν ήταν αντικείμενο συνένεση. Αναφέρατε κύριε Μπαρνιέ το ζήτημα των λαθασμένων συμβουλών. Συμφωνήσαμε πως είναι λογικό να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο. Το θέμα δεν είναι ο ορισμός ε, και οι δομές για να εμποδιστούν αυτές οι λανθασμένες συμβουλές. Οπωσδήποτε αυτά ανήκουν στην οδηγία ΜΥΦΙΤ. Αλλά εάν μια επιχείρηση αποδεδειγμένα δίνει λανθασμένες συμβουλές και μετά έχει χρεοκοπήσει και δεν μπορεί να έχει ευθύνη, τότε δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και αυτοί ε, κατά συνέπεια χρεοκοπήσει δεν προστατεύονται. και αυτό το δείξαμε νομίζω στη διαβούλευση που έγινε στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων και σας παρακαλώ κύριε Μπαργή να επανεξετάσετε την αρνητική σας στάση. Επίσης το θέμα των ε, usage θα μας απασχολήσει ξανά αυτό το ζήτημα. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θεωρώ βασικό είναι πως ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ψηφία που μπλοκάρει στο Συμβούλιο και εκεί πέρα ανήκει και η γερμανική κυβέρνηση και θα πρέπει να σκεφτεί εάν θέλει να συνεχίσει να μπλοκάρει. Χρειαζόμαστε αυτή την ε, προστασία. Δεν έχουν πλέον άλλη κατανόηση οι πολίτες για τη μη προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Περνάμε στο κομμάτι και Πρώτος λοιπόν είναι ο κύριος Γκαμάλιστα, ο Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τον επίτροπο. Συχνά λέμε ότι αυτά τα μέτρα οφείλονται στον Μάντοφ. Αλλά η υπόθεση Μάντοφ θα δείτε ότι πολλέ φορές είχε πάει η υπηρεσία κινητών αξιών στο Μάντοφ χωρί να δει κάτι και ή είχε μέτρα που δεν χρησιμοποίησε. Αυτό που με ανησυχεί στην οδηγία είναι ότι δημιουργεί, ο, δημιουργείται ηθικός κίνδυνος. Δηλαδή, ε, παροτρύνονται οι επενδυτές να μην προσέχουν επαρκώς επενδύσεις τους. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Θέλω να ευχαριστήσω τις άλλες ομάδες που δέχθηκαν την τροπολογία μου για τη διαφάνεια. Είναι σημαντική να βλέπουν το κόστος του κανονισμού οι επενδυτές, αλλά καταλαβαίνουν και τι πληρώνουν για την αποζημίωση. Και να μην οδηγηθούν στο να πληρώσουν περισσότερο μια επένδυση. Αυτό που με ανησυχεί είναι η υψηλή αποζημίωση. Αυτό μπορεί να ισχύσει για το Λονδίνο, τη Φραγκφούρτη, το Παρίσι. Οι μικρές ωστόσο αγορές ε, φοβούνται την, την υπερβολική συγκέντρωση ποσών, ποσο, τέτοιων ποσοτήτων. Γι' αυτό το λόγο σε αυτό το σημείο θα απόσουμε, προσβλέπουμε σε μια ε, ωραία συζήτηση. Ο κύριος Μόλτσερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι χρηματαγορές ως ξέρετε ασχολούνται με προϊόντα περίπλοκα τα οποία γίνονται όλο και πιο ακατανόητα. Αυτό πλέον δεν αφορά μόνο τον μικρό επενδυτή όπως είδαμε στις ε, ΗΠΑ. Μια φορά και ευρωπαϊκές τράπεζες ε, ανταλλάσσουν ε, τεράστια ποσά μεταξύ τους τα οποία τελικά καταλήγουν να μην αξίζουν τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να περιοριστούν ορισμένε κερδοσκοπικέ πρακτικέ, όπως οι ακάλυπτες, όπως ξέρετε, ανοιχτέ πωλήσει και θα πρέπει να έχουμε και αυτό το σύστημα αποζημίωση των επενδυτών. Θεωρώ τώρα πως η οδηγία θα πρέπει να προσανατολιστεί περισσότερο στην προστασία των καταναλωτών και νομίζω πως οι αλλαγές που επέφερε ο εισηγητής στο κείμενο της Κομισιόν είναι πάρα πολύ θετικές, ειδικά όσον αφορά το διασυναριακό χαρακτήρα όπου πρέπει να υπάρχει μια προβλεψιμότητα και νομική ασφάλεια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, ένα κοινό επίπεδο προστασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κυρία Πρόεδρε. Για τον κύριο Μπόντιου καταρχήν θα ήθελα πολύ λακωνικά να εκφράσω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε. Βέβαια είναι διαφορετική η κατάσταση μεταξύ των αξιογράφων και των καταθέσεων αλλά εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε μια επαρκής χρηματοδότηση εγώ θα υποστήριζα την ευθυγράμμιση την οποία αναφέρει η κυρία Μπερές σε σχέση με το επίπεδο αποζημιώσεων, το κατόφλιο των αποζημίσεων για την επέκταση στους ΟΣΕΚΑ. Εγώ ξέρω το, τη θέση του Κοινοβουλίου για τα ζητήματα αυτά, αλλά παρόλα αυτά κύριε Γκοζές, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ενταχθούν εν καιρό, να ενταχθούν τουλάχιστον στο στη σφαίρα εφαρμογής τη οδηγίας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε οι μεν τους δε για το θέμα αυτό. Κύριε Γκοζές, πιστεύω επίσης ότι <clears throat> όλοι οι επενδυτέ θα πρέπει να βρίσκονται σε επίπεδο ισότητο. Σα ευχαριστώ που υποστηρίξατε την ανάγκη να υποστηριχθούν και να προστατευτούν οι επενδυτέ. Όπω είπε και ο κύριος Μέλσερ. Κυρία Περές, και εγώ τόνισα τη σημασία να σκεφτούμε όλα αυτά μέσα σε ένα γενικό πακέτο, να μην δούμε το κείμενο αυτό ε, μεμονωμένα. Και το μελλοντικό κείμενο σε σχέση με την ε, προστασία των αξιογράφων είναι μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν στην περίπτωση Μάντοφ. Ε, το θέμα τώρα των ασφαλιστικών συμβολέων, αυτό είναι μια επίσης πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχουν εδώ τεχνικά προβλήματα τα οποία θα προκύψουν από την ευθυγράμμιση των ασφαλιστικών συμβολέων. Και από την άλλη μεριά, το θέμα του υπερβολικού χρέους που έχουν συνάψει οι ορισμένες τοπικές και περιφερειακές αρχές και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε από κοινού το θέμα αυτό. Τέλος, κυρία Μπέρας, όπως και ο κύριος Γκίγκολτ, αναφέρατε το θέμα των κακών συμβουλών. Είναι θεμητό το ερώτημα αυτό. Θέλουμε να προστατέψουμε τους ανθρώπους, αλλά είναι αυτός ο σωστός νομικός τρόμος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα νομοτεχνικό θέμα που μπορεί να υπάρχουν εδώ διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν κύριε Γκίγκολτ να έχουμε μια εναρμονισμένη και συνεκτική ερμηνεία του τι σημαίνει κακή συμβουλή. Καταλαβαίνω βέβαια την επιμονή σας για το θέμα αυτό. Θα το μελετήσουμε στο φως της συζήτησης που συνεχίζεται σήμερα και εγώ κατέγραψα όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Ο εισηγητής μας για να κλείσει τη συζήτηση. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπορεί να μην το είπα στο ξεκίνημα. Πιστεύω ωστόσο πραγματικά στην ελεύθερη αγορά. Ο καθένας πρέπει να μπορεί να κάνει ελεύθερες επιλογές. Ταυτόχρονα, να το πω επίσης ευθέως, πιστεύω και στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται. Η οδηγία αυτή είναι σημαντική ακριβώς από αυτή την οπτική γωνία, με αυτή την αφετηρία. Συνάδελφοι, εσείς που με κατακρίνετε σε άλλα πλαίσια, θα έλεγα ότι είμαστε ακριβώς, έχουμε ακριβώς τις ίδιες θέσεις. Οι απλοί συνηθισμένοι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι πάνω κάτω μπορούν να κάνουν γαλήνη επένδυση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την, το μέλλον της Ευρώπης και για την χρηματοοικονομική αγορά. Μίλησε ο κύριος Μπανιέ για την ΟΣΕΚΑ. Μπορούμε να συζητήσουμε ε, για αυτό το θέμα, μπορούμε να συζητήσουμε για το 0,3% πάνω, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αλλά το Συμβούλιο θέλει ε, ναι, πολύ χαμηλότερους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Ίσως λοιπόν δεν είναι τόσο άνετη η κατάσταση. Κατέγραψε επίσης αυτά που αναφέρθηκαν για τους ΟΣΕΚΑ και την ΜΥΦΙΔ. Νομίζω ότι θα βρούμε μια συμφωνία από αυτού. Σε ό,τι αφορά τώρα το λεγόμενο bad advice, την κακή αρνητική συμβουλευτική, κατά άποψή μου είναι πολύ σημαντικό σημείο για τους επενδυτές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και τέλος, Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο τον και όλους τους συναδέλφους, ε, τους κοιόδους για την πολύ χρήσιμη ε, συνεργασία τους στο δύσκολο αυτό θέμα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται τώρα η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το οποίο είναι η έκθεση Κοέλιο για τον Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Μεγάλων Πληροφοριακών Συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Και πριν ξεκινήσει η συζήτηση να πω πως ε, αναμέναμε την κυρία Μάλεμστρομ να είναι εδώ, αλλά καταλαβαίνω πως υπάρχει ένα πρόβλημα με την πτήση.